Τώρα, στην ημερησία διάταξη έχουμε την κοινή συζήτηση σχετικά με τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Έκθεση Μαρινέσκου για την υλοποίηση του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού και την έκθεση Σασόλη, αεροδρόμια, διαχείριση της ενέργειας κυκλοφορίας και υπηρεσίες αεροπλοείας. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή κύριο Μαρινέσκου για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Γύρω στις 26.000 ε, πτήσεις το χρόνο, μισό εκατομμύριο επιβάτες. Τα εργασίες, χιλιάδες θέσεις εργασίας στις αεροπορικές εταιρείες, 100.000 εργαζόμενοι τον ε, έλεγχο αέρες κυκλοφορίες, ε, μπλοκαρισμένοι δρόμοι. Γιατί, γιατί υπάρχουν μονοπόλια των κρατών μελών στον έλεγχο αέρες κυκλοφορίες. Και είναι το τελευταίο τέτοιο μονοπόλιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δούμε τις αερομεταφορές. Όταν λοιπόν συντάσσουμε νομοθεσία πρέπει να λάβουμε υπόψη όλου του ενδιαφερόμενου ε, ανθρώπου, εταιρείε, διοίκηση. Αυτή τη φορά λοιπόν θα κερδίσουμε μια αρχιτεκτονική η οποία θα βασίζεται στην αποτελεσματικότητα και όχι στα σύνορα και τη δρομολόγια. Το αποτέλεσμα λοιπόν θα είναι 15 λεπτά λιγότερα σε κάθε πτήση δύο ωρών. Άρα λιγότερα καύσιμα, λιγότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, χαμηλότερο κόστος και χαμηλότερες τιμές για τους επιβάτες. Αυτός ήταν ο στόχος ε, του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού 1 και δύο και δύο συν. Η εφαρμογή λοιπόν των κανονισμών αυτών Επέφερε κάποια πρόοδο, είχαμε κάποια σχέδια απόδοσης, φορείς αξιολόγησης της απόδοσης, λιγότερες καθυστερήσεις ε, και το κόστος των ε, εταιριών όμως και των επιβατών δεν έπεσε γιατί δεν έχει αναδιαμορφωθεί ο αέριος χώρος, ε, δεν υπάρχουν μπλοκ ενεργείου χώρου και δεν υπάρχει κάποια πρόοδος για πολιτικούς λόγους τα κράτη και τα συνδικάτα και οι διοικήσεις προσπαθούν να διατηρήσουν τα προνόμια τους, φοβούνται αδικαιολόγητα ότι θα χάσουν ε, θέσεις εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει τεράστια χρήματα και ο κλάδος επίσης σε νέα τεχνολογία και τα πρώτα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά και θα είναι κρίμα ή εφαρμογή να γίνει με την τωρινή αρχιτεκτονική. Θα έχουμε σημαντική σπατάλη ε, δημόσιου χρήματος και δεν θα έχουμε τα προσδοκόμενα ωφέλη. Έχουμε λοιπόν κάποιες προτάσεις ε, από τον κανονισμό. Θα υπάρχει μια διαχείριση από έναν διαχειριστή, μια κατανομή ανάλογα με την αποτελεσματικότητα, η δυνατότητα επανεξέτασης του εναέριου χώρου, και βεβαίως ε, θα υπάρχει η δυνατότητα και η και οι εθνικές εποπτικές αρχές να ε, έχουν έναν ισχυρότερο ρόλο βεβαίως ε, κάποια πράγματα καταψηφίστηκαν στην Επιτροπή Μεταφορών. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πρόβλημα με αυτή την πρόταση, απλά προτείνουμε πράγματα που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ειδικά όσοι ωφελούνται από αυτή την διαδικασία. Οι επιβάτες δηλαδή, αυτό το οποίο α, αυτοί οι οποίοι δεν το θέλουν, γιατί δεν το θέλουν. Οι διοικήσεις των κρατών μελών και τα κράτη-μέλη ασχολούνται όχι με την εξυπηρέτηση των επιβατών, αλλά με τις διοικήσεις και τους, τα, τα συνδικάτα των εργαζομένων. Μα κάποια στιγμή πρέπει να λάβουμε υπόψη και τους χρήστες. Λυπάμαι ειλικρινά για το ότι δύο προεδρίες, η Λιθουανική και η Ελληνική, δεν μπόρεσαν καν να ξεκινήσουν τι συζητήσεις στο Συμβούλιο. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει πως τα κράτη-μέλη ξέρουν πως δεν έχουν τίποτα να αντιτάξουν στις ε, προτάσεις μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τα 4 λεπτά, κύριε Σασόλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ καταρχήν τους και τις που συνεργάστηκαν με πολύ επικοδομητικό τρόπο για τη σύνταξη αυτού του κειμένου για τον κανονισμό για τα αεροδρόμια, τη διαχείριση της ενέργειας κυκλοφορίας και υπηρεσίε αεροπλοεία και του Ευρωπαϊκού χώρου. όπω ξέρετε ανήκουν σε μία δεσμή μέτρων που παρουσίασε τον Ιούνιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο στόχο είναι να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα του οργανισμού διαχείριση των αερίου χώρου μέσω μεταρρύθμιση του τομέα τη παροχή υπηρεσιών αεροπλοεία. Το κείμενο με τον ενίο Ευρωπαϊκό Ουρανό είναι πολύ ε, πλήρε, δεδομένε τη επίπτωση στα διάφορα κράτη-μέλη, είναι πολύ ευρύ και αντιμετωπίζει τα πιο επίμαχα θέματα. Καταρχήν, ε, την, έλλειψη, την ελλειπή αποτελεσματικότητα στην παροχή υπηρεσιών αεροπλοεία. Ε, δεύτερον, τον κατακαιρματισμό των συστημάτων διαχείριση τη ενέργεια κυκλοφορία. Ο κανονισμό αντιμετωπίζει το θέμα που έχει να κάνει με την ενεργία ασφάλεια και τις αρμοδιότητες ε, του οργανισμού. Θέλουμε να έχουμε ένα ε, ομοιόμορφο επίπεδο της ασφάλειας της αεροπλοείας στην Ευρώπη. Πρόκειται για ένα πολύ τεχνικό κείμενα που ρυθμίζει και το θέμα της διακυβέρνησης. Το πρώτο τμήμα του κειμένου έχει ως ε, θέμα την προσαρμογή στους νέους κανόνες ε, του ευρωπαϊκού, του ενίου ευρωπαϊκού ουρανού, ενώ το δεύτερο τμήμα αντιμετωπίζει το θέμα της μεταρρύθμισης ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση της υπηρεσίας. Για τις τεχνικές πτυχές του οργανισμού άκουσα διαφερόμενα μέρη, την Κομισιόν, και υπήρξε ομοφωνία για το κείμενο που παρουσιάστηκε. Ο κανονισμός θα εφαρμοστεί στο σχεδιασμό, στην παραγωγή, στις επιχειρησιακές στοιχές ε, των ερνευτικών προϊόντων. Συμπεριλαμβάνονται εκεί και οι υπηρεσίες αεροπλοείας και η διαχείριση της ενέργειας κυκλοφορίας, αλλά και τα πιστοποιητικά των πιλότων. Και εδώ στόχος είναι να διατηρήσουμε ένα υψηλό και ομοιόμορφο επίπεδο ασφάλειας διαφέρει τώρα το θέμα της διακυβέρνησης ε, του οργανισμού που ρυθμίζεται στο δεύτερο τμήμα του κανονισμού κομισιών παρουσίασε μια καινοτόμο πρόταση προβλέπεται μεταρρύθμιση του ίδιου του οργανισμού και δυνάμει μια ανακατανομής αρμοδιοτήτων καθορίζοντα ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας η ΆΖΕ θα επικεντρωθεί ε, στην εποπτεία της ε, ε, των τεχνικών ε, κανονισμών της ασφάλειας, ε, Control για τις επιχειρησιακά καθήκοντα. Και αυτή η μεταρρύθμιση ήταν προφανής από την αρχή, καθώς η Κομισιόν ήθελε να τροποποιήσει και το ίδιο το όνομα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού να ήθελε να μιλήσει για αεροπορικό οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν έδειξε ότι ήθελε να ακολουθήσει το παράδειγμα της Αμερικανικής κυβέρνησης ήθελε η Κομισιόν ε, να θέσει σε εφαρμογή τη Διοργανική Συμφωνία του Ιουλίου του 2012. Επομένω, ε, τα τρία θεσμικά όργανα βρήκαν μια συμφωνία για μια κοινή προσέγγιση για τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς που αν και δεν είναι νομικά δεσμευτικό, βασίζεται σε μια προσέγγιση ένα περίπτωση και σημειώνει πρόοδο σε πάρα πολλέ πτυχέ. η επιλογή της έδρας, διακυβέρνηση, λειτουργία, χρήση των πόρων ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας είναι ένας από τους πιο σημαντικούς οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό το λόγο ο Διευθυντής θα πρέπει να λογοδοτεί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Αρμόδια Επιτροπή για τις Μεταφορές σε σχέση με τις δραστηριότητες και τον προγραμματισμό του οργανισμού. Συνεχίζει να εξελίσσεται ο κλάδος της αεροπλοείας στην Ένωση. Ξέρετε ότι ο το στόχος είναι η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα σε έναν κόσμο όπου φυσικά συνεχώς αυξάνεται ο ρυθμός των πτήσεων. Θα είναι σημαντικό να κατανοήσουμε το ρόλο της Ευρώπης. Τα κράτη-μέλη ε, δεν μπορούν πλέον να συναγωνιστούν με τις μεγάλες χώρες των άλλων επίρων και μόνο μία όλο και πιο εξορθολογισμένη διαχείριση θα μπορέσει να μας οδηγήσει σε μεγαλύτερη ασφάλεια και σε ανταγωνιστική ικανότητα. Θα μειωθεί αμέσω το κόστο, των εισιτηρίων, θα ενισχυθεί η ασφάλεια, θα έχουμε μείωση του κετεκερματισμού, του ελέγχου, μείωση ε, της χρήσης των καυσίμων, λιγότερη ρήπανση, λιγότερες καθυστερήσει, μικρότερες καθυστερήσει στι πτήσει. Επομένως, είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση που θα μπορούσε μάλλον να είναι και πολύ ενδιαφέρουσα για την ανάκαμψη της οικονομίας μας. Θέλω να κάνω μια τεχνική διευκρίνηση, Πρόεδρε, επειδή υπάρχει ένα λάθος ε, επικοινωνίας της γραμματείας, δεν έχουν ε, μπει στο κείμενο δύο τροπολογίες για αύριο, η 43 και η 44, που ψηφίστηκαν στην Επιτροπή στις 30 Ιανουαρίου. Δεν ε, θα είναι δυνατόν λοιπόν να τροποποιηθεί το κείμενο που θα παρουσιαστεί εδώ, επειδή δεν ήταν μάλλον συγγνώμη δυνατόν να τροπεί το κείμενο, θα μπουν δύο αυτές τροπολογίες στον ευριανό κατάλογο. Ευχαριστώ, η Επίτροπος Ρέντινγκ. Αυτή η πρωτοβουλία για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα στον χώρο της εναέρειας κυκλοφορίας. Αυτή τη στιγμή είναι κατακαιρεμανισμένο το σύστημα και έχει πάρα πολλές καθυστερήσεις. Δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιτήρηση. Είναι υπεπαλαιωμένη η τεχνολογία και είναι και πολύ πιο δαπανηρό από τα συγκρίσιμα αλλού. Άρα λοιπόν με το project αυτό κάναμε το πρώτο βήμα για να αντιμετωπίζουμε τα θέματα αυτά. Δηλαδή πραγματική παρακολούθηση, εξυγχρονισμός μέσω τεχνολογίας και για πρώτη φορά στην ιστορία της αερο... αεροπλοείας μειώσαμε την αύξηση του κόστους. Αν λοιπόν τα κάναμε όλα αυτά θα μου πείτε Αφού είναι τόσο καταπληκτικά, γιατί να σας καταθέσω νέα πρόταση. Η απάντηση είναι πως αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην αφετηρία μιας μακριάς διαδρομής και ενώ έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος δεν είμαστε πουθενά κοντά στους στόχους μας. Είναι, είναι δύο πρωτοβουλία που δεν πρόκειται να παρουσιάσει κάποια νέα πολιτική, αλλά θα μας, επιτρέψει να πάμε στην επόμενη φάση υλοποίησης υφιστάμενων πολιτικών για να κατακτήσουμε αυτά τα οποία χρειαζόμαστε. Άρα λοιπόν έτσι γίνεται η ασφάλεια και η παρακολούθηση αντικείμενο μιας ανεξάρτητης εποπτικής αρχής. Και παρόλο που ακούγεται αξιοσημείωτο, ακόμα έχουμε κάποιους, ε, ε, κάποιες περιοχές όπου πολλές φορές αυτές οι αρχές όχι μόνο επιβλέπονται από όσους επιβλέπουν αλλά στελεχώνονται και από όσους επιβλέπουν. Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι συνταγή ε, για ε, μια παρακολούθηση στεναρή του θέματος ασφάλειας. Τώρα για, του ε, τους ελέγχους και την περιοχή ελέγχων, ελέγχων εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θέλουμε μεγαλύτερη διαφάνεια, Θέλουμε να έχουμε ε, εναέριες υπηρεσίες οι οποίες δεν ακολουθούν σήμερα ακόμα την νομοθεσία περί κρατικών προμηθειών και αυτό δημιουργεί κάποιες ε, αθέμητες πρακτικές. Η πρόταση λοιπόν δίνει ε, μία προώθηση σε αυτά τα FAB, τα λειτουργικά τμήματα ενιαίου εναέριου χώρου, με συγχωρείτε, και η διαδικασία λήψη αποφάσεων για τις αποδόσεις είναι εξορθολογισμένη και πιο ανεξάρτητη. Σχετικά με τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου Καταλαβαίνω πως σε κάποια κράτη η ιδέα αυτής της αρχής της ανεξάρτητης που θα επιβλέπει είναι δύσκολη. Αν όμως οι εθνικές αρχές δεν δώσουν τα κονδύλια και την ανεξαρτησία που χρειάζεται, δεν θα φτάσουμε ποτέ να έχουμε αρκετή ασφάλεια στον ενιαίο ε, ευρωπαϊκό ουρανό. Έχουμε αντιμετωπίσει μεγάλα κενά στην επιβλέψη, τα οποία θα πρέπει να ε, διορθώσουμε πριν έχουμε ατυχήματα. Και έχουμε και με κάποιες, ε, ε κάποιες ανησυχίες για κάποιες διατάξεις ε, που καταργούν τις διακρίσεις τους παρόχους υπηρεσιών τα, τους ANSP. Ε, νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό τα αντικειμενικά κριτήρια ε, δεν ε, δικαιολογούνται αρκετά, δεν τεκμηριώνονται και κάπου εξαλείφονται και οι διακρίσεις. Εμείς θέλουμε να αποτελεί βασικό κοινωνισμό που θα βοηθήσει να ξεπερασούν τα προβλήματα και είναι πολύ λίγα τα σημεία στα οποία εμείς δεν συμμεριζόμαστε τα όσα είπε η Επιτροπή Τραν. Για τις κατεξουσιοδότηση πράξη. εμείς θεωρούμε πως το κείμενο θα πρέπει να ακολουθήσει τη συνήθεια τακτική για τις κατεξουσιοδότηση πράξη και να μην εισάγει νέες διεκδικήσεις παρόλο που εμείς είπαμε οι εμπειρογνώμονες και οι ομάδες των εμπειρογνωμόνων που προτάθηκαν μπορούν να γίνουν δεκτά. Επίσης θέλουμε να διατηρηθούν μια αξιολόγηση στο τέλος της θητείας του ε, εκτελεστικού διευθυντή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό αν πρόκειται κανείς να επαναδιοριστεί. Θα κλείσω ευχαριστώντας και πάλι το Κοινοβούλιο για τη στήριξη που προσφέρει και πιστεύουμε πως η επιτυχής πρώτη ανάγνωση ε, θα πιέσει το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη να κάνουν αυτό το οποίο πρέπει. Ευχαριστώ. Τώρα. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Ρικέ από το ΕΛΚΕ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τους δύο ε, για ένα πολύ δύσκολο έργο, ε, για ένα θέμα που δυσκολεύεται να προχωρήσει. Τα θέματα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκος προς τις διαδικασίες ε, και προς τους πρωταγωνιστές. Υπάρχουν πολύ μεγάλα θέματα περιβαλλοντικά και οικονομικά. Όλες ε, οι προβλέψεις δείχνουν ότι θα αυξηθεί τα επόμενα έτη η ενέργεια κυκλοφορία, όμως δυστυχώς δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι και υπάρχει μεγάλος κατακαιρματισμός ε, στον ενέργειο χώρο και αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει συμφόρηση του ενέργειου χώρου με, εσωτερικά, με εσωτερικό κόστος, αντίκτυπο στο περιβάλλον ε, και θα έχουμε υπερβολικά και κατανάλωση καυσίμων και η ποιότητα ε, για την παροχή υπηρεσιών ε, θα επιδεινωθεί. Ε, ο νέος Ευρωπαϊκός Ουρανός ε, θα έχει θετικό αντίκτυπο για την ανάπτυξη της απασχόλησης και της οικονομίας στην Ευρώπη. Αναφέρθηκε ο κύριος Μαρινέσκου στη σημασία του κλάδου για την οικονομία και ε, για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Έχουμε κάποιες εταιρείες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Θα πρέπει να υπερασπίσουμε πιο οικονομικά με ταξίδια και θα πρέπει να υπάρχει διαλειτουργικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να βελτιωθεί χρησιμοποιώντας και το σύστημα ΣΕΖΑΡ παράλληλα με τον Ευρωπαϊκό Ουρανό παρά τις πραγματικές δυσκολίες ε, μπροστά σε εθνικές εμπλοκές ε, τελικά ε, φτάσαμε στο να έχουμε πραγματική ολοκλήρωση του ενίου ευρωπαϊκού ουρανού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δανέλης για τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες για 4 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Λίγο πριν τις ευρωεκλογέ και μάλιστα με διαβρινόμενο τον ευρωσκεπτικισμό, καλούμαστε να πείσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες πως η Ένωση είναι χρήσιμη στους πολίτες της και για τα μικρά αλλά και για τα μεγάλα. η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά στις αερομεταφορές τα τελευταία 20 χρόνια έχει καταστήσει τις πτήσεις προσιτές σε εκατομμύρια νέους επιβάτες αλλά η αυξανόμενη κίνηση ασκεί τεράστιες πιέσεις στη διαχείριση της εναέρειας κυκλοφορίας και όσο κλιμακώνεται η κίνηση θα έχουμε ολοένα και περισσότερες καθυστερήσεις λιγότερες και ακριβότερες πτήσεις αλλά και ερωτηματικά σχετικά με την πτυτική ασφάλεια. οι υπηρεσίε και κυκλοφορία δεν είναι προετοιμασμένε για τον 21ο αιώνα και ο συνδυασμό ασφαλών και φτηνών πτήσεων χωρί καθυστερήσει έχει δυστυχώ ημερομηνία λήξη. με την με την πρόφαση της εθνικής κυριαρχίας και της επικουρικότητας ο έλεγχος της εναέρειας κυκλοφορίας παραμένει εξ ολοκλήρου εθνική υπόθεση δέσμια στερεοτύπων ιδεολειψιών αλλά και συμφερόντων. για τον επιβάτη και για τις αεροπορικές εταιρείες της ένωσης η σημερινή κατάσταση των 38 διαφορετικών και ασύμβατων συστημάτων αεροναυτιλίας αλλά και των 60 διαφορετικών κέντρων ελέγχου είναι απαράδεκτα επιζήμια και φυσικά αυτό δεν έχει να κάνει με το αν ο πάροχος των υπηρεσιών είναι το δημόσιο ή κάποιος ιδιώτης. οι ηνωμένε πολιτείε τις παρέχουν δημόσια όπως και εμείς αλλά με ένα πάροχο αντί για τους 38 και εν τέλει με το μισό κόστος. Ας μην μας διαφεύγει όμως ότι η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών αεροδρομίων έναντι εκείνων της ανατολής δέχεται διαρκώς πίεση οι αλλαγές που χρειάζονται είναι οργανωτικές και δεν αφορούν την επάρκεια και την ικανότητα των στελεχών. αποτελεί επίτευγμα των υπηρεσιών αέρης κυκλοφορίας το ότι η μεγάλη αύξηση της κίνησης τα τελευταία 20 χρόνια πραγματοποιήθηκε με δεδομένη την ύψιστη εγγύηση ασφάλειας που γνωρίζουμε και βεβαίως απαιτούμε όταν πετάμε στην ευρώπη. αλλά για να κάνουμε το επόμενο βήμα πρέπει να προχωρήσουμε στον εξορθολογισμό δηλαδή επιτέλους στην υλοποίηση του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. μόνο έτσι θα ελαχιστοποιήσουμε τις διανυόμενες αποστάσεις με επακόλουθα τη μείωση της διάρκειας των ταξιδιών και της κατανάλωσης καυσίμων. αυτό θα σημάνει μείωση του περιβαλλοντικού κόστους αλλά και του οικονομικού κόστους για εταιρείε και για επιβάτες. με την έκθεση ενδυναμώνουμε το μηχανισμό επιδόσεων ώστε τα κράτη μέλη να συμμορφώνονται στους στόχους που τίθενται από την ευρωπαϊκή επιτροπή ισχυροποιούμε την εθνική εποπτεία δημιουργούμε προϋποθέσεις διαφάνειας στην παροχή των υποστηρικτικών υπηρεσιών και φέρνουμε για πρώτη φορά τον ανθρώπινο παράγοντα στο κέντρο του ενιαίου ουρανού. Ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός είναι ένα στίχημα. Ένα στίχημα ουσίας αλλά και συμβολισμού για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπροστά στις κοντόφθαλμες κολυσιεργίες του Συμβουλίου, το Κοινοβούλιο πρέπει αύριο να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα κλείνοντας θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τους εισηγητές για την πολύ καλή έκθεση και την άψογη συνεργασία που είχαμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ομάδα των φιλελεύθερων. Ο κύριος Μπένιον για δύο λεπτά. <coughs> Thank you, Chair, and thank you. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τον εισηγητή και τους συναδέλφους για τη δουλειά που έκαναν. Εγώ δεν θα πω ότι χρειαζόμαστε τώρα τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, τον χρειαζόμασταν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχω απογοητευτεί από την έλλειψη πολιτική βούληση από τα κράτη-μέλη για να υλοποιηθεί, αλλά χαίρομαι για το ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου στηρίζει τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Ναι, ναι, το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει περισσότερη Ευρώπη, παρά το ότι οι συντηρητικοί μα ε, σκέφτονται να βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κατακαιρματισμό του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου υπολογίζεται πω κοστίζει πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Κοστίζει θέσεις εργασία και αυξάνει τις εκπομπέ δεξιού του άνθρακα χωρίς να υπάρχει λόγος. Χρειάζεται πιο αποτελεσματικός εναέριος χώρος για να μην υπάρχει ε, κίνηση γύρω από τα αεροδρόμια και να ανταποκριθούμε στα ζητήματα του περιβάλλοντος. Επίσης θα πρέπει να γίνουν τώρα οι σωστές προσπάθειες. Ε, όμως είμαι πραγματικά απογοητευμένος για το ότι έχει παίξει ρόλο η εθνική πολιτική σκηνή σε ένα ζήτημα το οποίο υποτίθεται πως αφορά την ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Μα δεν υπάρχει καθόλου κοινή λογική. Με ποια λογική εξαιρέθηκε το Γιβραλτάρ. Η νομοθεσία αφορά τον ουρανό, τον έλεγχο αέρη κυκλοφορία και τη συνεργασία των ελεγκτών. Οι ελεγκτέ του αεροδρομίου του κ. δεν δουλεύουν μόνοι του, είναι σε επαφή συνεχώ με του Ισπανού συναδέλφου στη Σεβίλη. Γιατί λοιπόν κάποιοι συνάδελφοι θέλουν να εμποδίσουν αυτή την συνεργασία, γιατί να απομονώσουν το Γιβραλτάρ. Οι φιλελεύθεροι αύριο θα καταψηφίσουν όλες τις, τρομο... τις ε, τροπολογίες που αποκλείουν το Γιβραλτάρ και θα αποδείξουμε έτσι την δέσμευσή μας για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό και ίσως να χρειαστεί μάλιστα να αποσχούμε. Εάν και υπενθυμίζω εδώ πέρα πως το Γιβλατάρ είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκλειστεί από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Σας ζητώ λοιπόν να υποστηρίξετε την πρόταση της Κομισιόν που ήταν να συμπεριληφθεί το Γιβραλτάρ. Σας ζητώ να, ψηφί, να καταψηφίσετε την τροπολογία 27. Σας ευχαριστώ. Εξ ονόματος των Πρασίνων, η κυρία Λίχτενμπέργκερ έχει το λόγο. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε. Επί της αρχής είναι μια συναρπαστική ιδέα ο ενιαίος ουρανός, αλλά δυστυχώς ε, δεν μπορέσαμε να το περάσουμε γιατί είχαν αντιρρήσει τα κράτη-μέλη. Γιατί, γιατί το θεώρησαν κάτι το οποίο ε, μπορούν να εμποδίσουν γιατί ο εναέριος χώρος τους είναι δικός τους και κανένας άλλος δεν επιτρέπεται να κοιτάει τι γίνεται εκεί μέσα. Αυτή ήταν λίγο πολύ αιτιολογία για το ότι η εφαρμογή των λειτουργικών ε, μπλοκ εναέριου χώρου ε, δεν μπορεί να εφαρμοστεί όπως τα πρότεινε η Κομισιόν. Παρ' όλα αυτά υπήρξε κάποια πρόοδος. Υπάρχει σήμερα καλύτερη συνεργασία, καλύτερη οργάνωση οι καθυστερήσεις ε, πραγματικά έχουν μειωθεί. Τα δρομολόγια έχουν γίνει συντομότερα, αυτό οφείλεται και σε άλλα μέτρα βεβαίως. Ε, τα πεδία βολής είναι κάπως λιγότερα και οι απαγορευμένες ζώνες για στρατιωτικούς λόγους. Επίσης βεβαίως στο ζήτημα του διαχωρισμού έχει πάει κάπως μακριά η Κομισιόν, κάτι το οποίο απέρριψε η Επιτροπή Μεταφορών. Εγώ θα το διέγραφα τελείως γιατί είναι καθαρά ιδεολογικό το ζήτημα, δεν έχει ουδεμία σχέση με το ζήτημα. Αφορά τον διαχωρισμό των υπηρεσιών, κάτι το οποίο νομίζω πρέπει να το δούμε ανά κράτος μέλος. Πράξη κατεξιοδότηση τώρα τελευταία λέξη. Είναι μανία αυτή της Κομισιόν. Ε, βλέπω πως προσπαθείτε από την πίσω πόρτα να παρακάμψει το δημοκρατικό έλεγχο. Σας ευχαριστούμε. Εξ ονόματος του ECR, Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές, για 1,5 λεπτό, κυρία Φώστερ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν από 12 μήνες με μια δική μου έκθεση πρωτοβουλίας για την εφαρμογή του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού, είδα ότι είχα την ιδιαίτερη υποστήριξη των συναδέλφων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ζητούσα στην έκθεση αυτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματικά να συνειδητοποιήσουν πώ έχει κατάσταση. Επομένω, δεν μπορώ και παρά να χαιρετήσω την πρόταση αυτή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαι σαφώ υπέρ των βασικών στόχων της, του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού, καθώ επίση και υπέρ των τεχνικών στόχων του κ. Σάσολη. Υπάρχουν όμω κάποιε ανησυχίε όσον αφορά την έκθεση του κυρίου Μαρινέσκου. Δεν μπορούμε να δεχθούμε τη συγχώνευση εθνικών εποπτικών αρχών και εθνικών αεροπορικών αρχών στην ίδια αντότητα. Θα προκύψουν ζητήματα νομική φύση σε πολλά κράτη-μέλη, ιδίω στον Ηνωμένο Βασίλειο, που υπάρχουν πάρα πολλέ νομοθετικέ πράξει και οι οποίε θα πρέπει να τροποποιηθούν άνευ λόγου και αιτία. Δεύτερον, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την περαιτέρω ανεξαρτητοποίηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλεια τη Αεροπορία. Παρ' όλα αυτά πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είμαστε και πιο προσεκτικοί. Θα πρέπει να διευθυνθεί και το ζήτημα του, Γιβραλτά, του Γιβραλτάρ. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο ο προβλητικό τρόπο με τον οποίο έχουν αντιδράσει ορισμένοι Ισπανοί συνάδελφοι. Α μην ξεχνάμε ότι η συμφωνία του 2006 υπεγράφει από όλε τι πλευρέ. Α μην αποδεχθούμε αυτή τη στιγμή ένα κατακαιρματισμό του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Θεωρώ ότι η συμπεριφορά ορισμένων Ισπανών συναδέλφων είναι καθαρά παιδιάστικη και ουσιαστικά βάλει κατά μια πρωτοβουλία που δημιουργήσει χιλιάδε θέσεων εργασία, θα μειώσει τι τιμέ των αεροπορικών τιμών και επίση θα οδηγήσει σε μία μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Και ελπίζω συνάδελφοι από την ομάδα των Πρασίνων να με ακούνε. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν από του αδέλφου να στηρίξουν την πρόταση αυτή αύριο κατά την ψηφοφορία. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε. Εξ ονόματος της ε, ΓΚΟΕ, ο κύριος Κόλιτσεκ, για ένα λεπτό έχει το λόγο. Evropská komise, tak jak se blíží konec jejího mandátu, začíná připomínat sbor finišujících závodníků. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερα φιλελεύθερες ε, από οικονομικής πλευράς ε, προτάσεις. οι οποίε συμπεριλαμβάνονται και στην πρώτη πρόταση για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Η πρώτη αυτή πρόταση δεν έχει ακόμα αξιολογηθεί. Θεωρώ λοιπόν ότι προχωράμε αυτή τη στιγμή πάρα πολύ γρήγορα με την πρόταση SES 2+. Ο εισηγητή νομίζω ότι πολύ αφελώ υποστηρίζει την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορεί οι αεροπορικέ εταιρείε να βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με την κατάσταση τη διαχείριση ενιαία κυκλοφορία. Οι εθνικές αεροπορικές αρχές πολιτικής αεροπορίας ήδη συνεργάζονται πάρα πολύ καλά. Θεωρώ λοιπόν ότι η συγχώνευση που προτείνεται αυτή τη στιγμή ανάμεσα στις εθνικές υποπτικές αρχές και τις εθνικές αεροπορικές αρχές δεν είναι σωστή. Η ομάδα μου δεν πρόκειται να υποστηρίξει λοιπόν αυτή την πρόταση. Σας ευχαριστούμε. Τώρα το λόγο έχουν οι υπόλοιποι ομιλητέ. Πρώτος ο κύριος Ελκαντράουι για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι. Θέλω καταρχήν πρώτα να ξεκινήσω με τον εισηγητή και να αναφερθώ και στον κύριο Μαρινέσκου. Θέλω όλους αυτούς και τους συναδέλφους να τους ευχαριστήσω για την επικοδομητική συνεργασία. Ένας ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός είναι παλαιό όνειρο της Ευρωβουλής και κατά το παρελθόν κάναμε πολλά βήματα και διαβήματα προς την αυτή την κατεύθυνση. Είναι όμως ε, απόλυτη ανάγκη να βελτιωθούν τα πράγματα ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Είναι καλό και για την βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, εξοικονόμηση κόστους συνεπάγεται και λιγότερες καθυστερήσεις για τους επιβάτες και χαμηλότερες τιμές, πιο προσιτές τιμές και για το περιβάλλον είναι επίσης καλό, διότι θα εκλείονται μικρότεροι όγκοι ε, διοξιδίου του άνθρακα και θα καίγεται ε, λιγότερο καύσιμο. Είναι λοιπόν ένα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση, σίγουρα αυτό και το επιθυμούμε και θέλουμε να γίνει. Από αφήνιση και των ευθυνών και μέσα σε ένα πιο ορθολογικό πλαίσιο και ένα πιο αποτελεσματικό πλαίσιο. Και οι προλαλήσαντες και οι σε ήδη τα προανέφεραν αυτά. Δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι δεν θα υποστηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν έχουμε και την, ε, την πρόταση μιας υποχρεωτικής, ενός υποχρεωτικού διαχωρισμού υπηρεσιών. Το βασικό κείμενο είναι αποδεκτό, αλλά καταθέσαμε τροπολογία που θα ψηφιστούν αύριο. Παραμένουν πολλά όμω που πρέπει να γίνουν και πολλά εξαρτώνται από τα αποτελέσματα επιτόπου και από την υλοποίηση και εφαρμογή στα κράτη-μέλη. Το είδαμε αυτό και με το SAS2 ε, Single ε, European Skies SES. Ε, e θα ήθελα να αναφερθώ στην Επιτροπή που θα έπρεπε να επικεντρωθεί στα πρακτικά προβλήματα και για το πώς θα επιμεριστούν τα κόστη και τα έσοδα όσον αφορά τις εταιρείε. Ε, όταν θέλουμε να υπάρχει αποτελεσματικότερο πλαίσιο πρέπει τότε να έχουμε και ένα καταστατικό για τους υπαλλήλου ώστε σε αυτό τον τομέα να υπάρχει ένα θετικό μέλλον ως προοπτική. Σας ευχαριστούμε ο κύριος Βλάζακ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η ιδέα αυτή της πιο αποτελεσματικής χρήσης του ευρωπαϊκού χώρου, εναέριου χώρου, είναι κάτι που υποστηρίζαμε. Όμως στο SE, ε, Single European Sky Plus υπάρχουν κάποια προβλήματα. Είναι προβληματική πρόταση. Σε λάθος χρονική στιγμή και συγκυρία υποβάλλεται η πρόταση. Προτού μπορέσει να αξιολογηθεί η περίοδος αναφοράς για τον ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό 1 και που SES ε, 2 e που θα λύγει το 2014 έχουμε μια δραματικής μορφής πρόταση που δεν μπορώ να υποστηρίξω. Θα υπάρξουν αλλαγές όσον αφορά τη διαχείριση της δομής του εναέριου χώρου που οδηγεί σαφώς στην αποδυνάμωση της θέσης των κρατών μελών όσον αφορά την λήψη αποφάσεων ακριβώς σε θέματα που αφορούν τον ενιαίο ουρανό και επίσης ε, ε, εδώ σε σχέση με τα, κράτη-μέλη δημιουργούνται προβλήματα. Θετικό θα ήταν να αποσαφινιστούν πρώτα οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε και του, της Eurocontrol. Δεν μπορώ να υποστηρίξω λοιπόν αυτή την έκθεση. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Λιαρίκη για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Φοβάμαι ότι πίσω από τις ωραίες αυτές προθέσεις, ποετικές θα έλεγα, για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, κρύβεται τελικά ένα πολύ επικίνδυνο σχέδιο, το οποίο έχει ως στόχο να απελευθερώσει οικονομικά όλες τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρησιμοποιούνται διάφορα πολύ όμορφα λόγια, μια πολύ ευχάριστη διατύπωση, η οποία όμως τελικά θα οδηγήσει σε μια απορρίθμιση όλων των υπηρεσιών εποπτείας, που πραγματικά διοργανώνταν πάρα πολύ καλά από την Εθνική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Γαλλίας και από τις υπόλοιπες εθνικές αεροπορικές αρχές. Μιλάμε πραγματικά εδώ πέρα για μια διάλυση των εθνικών αυτών συστημάτων, όπου θα έχουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα πολύ πιο φτηνό, με λιγότερο προσωπικό, το οποίο θα υποπληρώνεται και που δυστυχώ θα οδηγήσει σε χαμηλό επίπεδο ασφάλειας για του ίδιου του επιβάτε, του αξιδιώτε, Στο όνομα λοιπόν τη ασφάλεια, τη ενέργεια κυκλοφορία, στο όνομα των επιβατών οι οποίοι θέλουν να μπορούν να ταξιδεύουν σε συνθήκες ασφάλειας, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να ξεφύγουμε από το επικίνδυνο αυτό σχέδιο. Δεν μπορούμε το, ο βασικός μας γνώμονας να είναι ο οικονομικός παράγοντας. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον οικονομικό παράγοντα ως βασικό επιχείρημα και να διακινδυνεύουμε τις ίδιες τις ζωές των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ταξιδεύουν. Γκέρλινγκ, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφοι. Βρίσκομαι σήμερα εδώ και νομίζω είμαι το μόνο μέλος που αντιπροσωπεύει το Γιβραλτάρ για να μιλήσω μόνο για αυτό το θέμα. Δεν ισχυρίζομαι ότι είμαι εμπειρογνώμονα για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, αλλά είμαι σε μια θέση όπου για δεύτερη φορά αυτούς τους μήνες πρέπει να σταθώ εδώ και να θέσω ερωτήματα σχετικά με το γιατί μέλη αυτού του σώματος επιχειρούν να κάνουν διακρίσεις κατά τη του, εκλογικής μου περιφέρειας στο Γιβραλτάρ. Δεν γνωρίζω τον κύριο Τεγκράντ Πασκουάλ που έχει προτείνει τι τροπολογίε 22, 23, 26 και 25, αλλά θα ήθελα να έχω μια συνομιλία μαζί του για να δω κατά πόσο πιστεύει ότι είναι αναγκαίο. Είναι επιτακτικό το Γιβραλτάρ να συμπεριληφθεί στην ενιαία αγορά τη αεροπορία μαζί με τι συνθήκε, σύμφωνα με τι συνθήκε. Ε, για την δική μου περιφέρεια στο Γιβραλτάρ φαίνεται να είναι συνεχώς ένα πρόβλημα μετά το άλλο. Συνεχώς καθυστερήσεις, ε, ε, τα προβλήματα με τα δικαιώματα των, επιβατών. Πότε θα σταματήσει αυτό. Θα ήθελα να άρουν αυτές τις τροπολογίες 22, 23, 25 και 26 και την 144 να ψηφίσουμε κατά των διακρίσεων. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στη δικασία Catch the Eye. Μπάνκι παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ο ενίος Ευρωπαϊκός Ουρανός η αναθεώρησή του και η πρόταση ε, για νομοθεσία θέτει κάποια σημαντικά ερωτήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει τη δήλωσή της και συμφωνώ απόλυτα, δηλαδή ότι το πλαίσιο ΣΕΣ θα πρέπει να αναδιατυπωθεί διότι δεν δουλεύει αποτελεσματικά μέχρι σήμερα. Η Επιτροπή έχει κάνει μια πρόταση, δυστυχώς αυτή δεν είναι απόλυτα σωστή, διότι δίνει πλεονέκτημα σε μεγαλύτερους φορείς και μειονεκτήματα σε μικρότερους φορείς, για παράδειγμα αυτού το περαιτέρω που λειτουργούν στην Ουγγαρία ε, για τον έλεγχο της ενεργής κυκλοφορίας, που είναι νέοι. Επίσης, οι υπηρεσίες έχουν ξεχωριστεί. Ε, μιλούμε για την ε, έννοια της ΣΕΣ 2 και πάμε σύμφωνα με αυτή την έννοια. Υπάρχουν κάποιοι μεγάλοι χειριστές που έχουν ένα πλεονέκτημα και θα ενισχυθούν και αυτό θα οδηγήσει σε περισσότερο κόστος. Ε, εισάγονται κάποιοι περιορισμοί στην αγορά που θα αποτελέσουν εμπόδιο στην ανταγωνισμό και νομίζω θα αποτελέσουν και κίνδυνο μακροπρόθεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ζουάμπ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Αντιπρόεδρε, καταρχήν πρώτα θα ήθελα τον συνάδελφο Μαρινέσκου και τους κοιόδης εισηγητές να ευχαριστήσω για την εξαιρετική δουλειά για την έκθεση για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Πιστεύω ότι ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός είναι ένα σημαντικό υπόδειγμα ως παράδειγμα πώς μπορούμε να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ευρωπαϊκή πρόσθετη αξία μέσω της συνεργασίας για πιο φιλοπεριβαλλοντικές ενέργειες μεταφορές και πιο προσιτές διασυνδέσεις στις ενέργειες μεταφορές. Αυτό το εγχείρημα ιδιαίτερα όσον αφορά την υλοποίησή του στα κράτη-μέλη θα πρέπει να το προαγάγουμε σίγουρα. Ως κάτοικος μιας μεθοριακής περιοχής με πολλές ε, τέτοιες, ε, ε, πολλούς τέτοιους δεσμούς γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει η υποδομή των αεροδρομίων και των εναερίων μεταφορών. Γι' αυτό πρέπει περισσότερα να επενδύσουμε η ενιοποίηση αυτού του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού να επιτευχθεί όχι μόνο με την επίτευξη των καλύτερων ας διασυνδέσεων αλλά και της καλύτερης ασφάλειας. Δυστυχώς εξακολουθούν αυτά να είναι θέματα εθνικά. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το Ευρωκοινοβούλιο εδώ να δώσει το παράδειγμα κάνοντας τα πρώτα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Σουάμπ. Στη συνέχεια ο κύριος Πικούλα παρακαλώ. Nastojanja komisije da se osigura siguran i visoko kvalitetan ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα πρέπει στον τομέα των αρμεταφορών να καταλήξουμε τελικά σε κάποια ταξίδια τα οποία θα είναι πιο φτηνά και πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Και βέβαια θα πρέπει να δημιουργήσουμε έναν ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, αλλά για αυτό το λόγο χρειαζόμαστε μία ισορροπημένη πρόταση. Νομίζω ότι θα πρέπει να θεωρήσουμε εκ νέου την πρόταση που έχουμε ενώπιό μας και να δούμε αν τελικά τίθεται ως προτεραιότητα η ίδια η ασφάλεια και αν η προτεραιότητα της ασφάλειας δεν βάλει κατά άλλων προτεραιοτήτων. Θα πρέπει να εξετάσουμε αν το εν λόγω σχέδιο θέτει να αμφιβόλο ή φέρνει σε πολύ δύσκολη κατάσταση κάποιες μικρές χώρες οι οποίες θα πρέπει να πιεστούν πάρα πολύ για να καταφέρουν ε, να ανταποκριθούν ε, στον καονισμό αυτό. Αναφέρομαι στις χώρες εκείνες που έχουν κάποια μικρά αεροδρόμια. Νομίζω ότι θα πρέπει να επεξεργαστούμε εκ νέου λίγο περισσότερο την πρόταση αυτή. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Στη συνέχεια Φερέρα. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Α είμαστε σαφεί. Η πρόθεση αυτού του πακέτου μέτρων είναι η απελευθερωποίηση και εμπορευματοποίηση τη διαχείριση του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου στην Ευρώπη. Να προχωρήσουμε για μια νέα μορφή εμπορίων. θέτοντα σε ευθυγράμμιση με τα συμφέροντα των μεγάλων εταιριών εναέριων μεταφορών τα πάντα. Αυτό είναι ο στόχο. Ο κατακαιρματισμό τη παροχή υπηρεσιών ε, ανταποκρίνεται στο, στο να ξεχαρβαλωθούν, να εναρμολογηθούν αυτές ε, οι επιχειρήσεις ε, που είναι ανταγωνιστικές. Εδώ όχι μόνο έχουμε το θέμα της ποιότητας αλλά και όλη την αλυσίδα ασφάλειας. Αμφισβητούνται και διακυβεύονται χιλιάδες θέσεις απασχόλησης ε, στις περιφερειακές χώρες. Διακυβεύεται η κυριαρχία, τα κυρίαρχα δικαιώματα των κρατών μελών και δεν υπάρχουν έτσι αυτές οι δυνατότητες διασφάλισης των πτυχών, της απασχόλησης, της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας των συνδέσεων και της ε, του δημόσιου χαρακτήρα αυτών των θεμάτων που θα έπρεπε πολύ καλύτερα να εξισωθούν και να αντιστοιχούνται γιατί διαφορετικά στην απελευθερώση αυτή έχουμε αρνητικές επιπτώσεις. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια κυρία Τίκαου παρακαλώ. Gracias. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να υπογραμμίσω την ε, σημασία της ε, εφαρμογής του ενίου ευρωπαϊκού ουρανού, διότι θα αυξήσει την ασφάλεια, θα μειώσει τις καθυστερήσεις. Αυτό θα βοηθήσει επίση και στην οικονομική μεγένθηση και στην απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, ιδιαίτερα την τόνωση των ε, ε, θέσεων απασχόληση. Βέβαια, η υλοποίηση του ΣΕΣ ε, εδώ οι παϊκοί ε, και οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να ενημερωθούν για τις κοινωνικές επιπτώσεις. Επίσης η ασφάλεια της αεροπορίας θα πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα. Δυστυχώς η υλοποίηση αυτής πρωτοβουλίας έχει καθυστέρηση σε ό,τι αφορά τις ε, επιδόσεις της ε, της, ε, του στόχους επιδόσεων. Αυτό θα έπρεπε να ήταν έτοιμο μέχρι το 2012 το Δεκέμβριο και θα είχε ως στόχο την ε, ενοποίηση των υπηρεσιών. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε κυρία Τικάου. Στη συνέχεια για ένα λεπτό η κυρία Λιπτσέβα παρακαλώ. Σα ευχαριστώ. Επιτροπή εισαγωγή ενός ε, ενιαίου νομοθετικού πλαισίου που θα συνενώνει τον ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό 1 και 2 δίνει προοπτικές αλλά για να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει να βρούμε τον χρόνο που οι χώρες θα είναι πραγματικά έτοιμες να αποδεχθούν αυτές τις προτάσεις ε, και τα κεκτημένα για να προχωρήσουν τον διαχωρισμό της διαχείρισης ε, των θεμάτων πτήσεων όπως υφίσταται στην πρόταση της Επιτροπής γιατί διαφορετικά θα επικεντρωθούν αυτές οι δραστηριότητες σε μεγαλύτερες εταιρείε. και αυτό θα έχει επιπτώσεις στις, στους υφιστάμενους εθνικούς μηχανισμούς γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και δεν θα πρέπει να κατηγορούμε τα κράτη-μέλη ότι δεν είναι ακόμα έτοιμα και όριμα να δεχθούν αυτή την τεχνολογία δεν μπορούν να επιτευχθούν όλα αυτά χωρίς μια μελέτη επιπτώσεων συμπεριλαμβανομένων και των κοινωνικών επιπτώσεων σε αυτή τη μελέτη επιπτώσεων. Μάλιστα, είμαστε όλοι υπέρ μεγαλύτερου ανταγωνισμού, περισσότερη ασφάλεια, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Σίγουρα. Όμω πρέπει να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τι θέσει απασχόληση και να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο σταθερότητα στο εθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια η Επίτροπος παρακαλώ θα λάβει τον λόγο. Πρόεδρε, ακούσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση εδώ σήμερα. Αντιλαμβάνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι κάποια τμήματα αυτή τη πρότασή τη μπορεί να δημιουργούν δυσκολίε ε, για επιμέρου εμπλεκόμενου. Όμω πρέπει να επικεντρωθούμε στα θετικά του συνολικού ε, συστήματο αν δεν υπάρξει ένα αναβαθμισμένο σύστημα όλοι θα υποστούν τις αρνητικές συνέπειες επιβάτες, ε, διαχειριστές όλοι. Όσον αφορά τις εποπτικές αρχές πιστεύουμε ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό πτυχή στην πρότασή μας και με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπω ότι υποστηρίζεται ευρέω αυτή η πρότασή μας. Επίσης το ίδιο ισχύει για τον εξορθολογισμό του θεσμικού πλαισίου και του ρυθμιστικού συστήματος. Από την άλλη πλευρά ο διαχωρισμός όσον αφορά τις υπηρεσίες εξακολουθεί να είναι σημαντικός όρος και προϋπόθεσης για να δημιουργηθεί ένα ισοδίκαιο πλαίσιο δραστηριότητας ε, για τις ε, επιχειρήσεις που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες. Και δεν θέλουμε να αποδυναμωθεί η πρότασή μας αυτή. Όσον αφορά την ιδέα του ε, EASA θα πρέπει να πιστοποιεί εθνικές αρχές, θεωρεί μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση αυτή την πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως θα είχε ευρύτερες επιπτώσεις και θα έπρεπε να γίνει μια σε βάθος μελέτη κάτι επιπτώσεων προτού γίνει δεκτό κάτι τέτοιο. Είναι πρόημο λοιπόν να γίνει δεκτό κάτι τέτοιο πρόταση. Επιφυλασσόμεθα να εξετάσουμε εν ευθέτω χρόνο περισσότερο την πρόταση αυτή σε βάθο. Εν συμπεράσματι, καλωσορίζουμε την θετική αντιμετώπιση του Ευρωκοινοβουλίου. Τώρα πρέπει επιτέλου να κινητοποιηθούμε και σε σχέση με το ευρωπαϊκό σύστημα ε, διαχείρισης πρέπει να αναβαθμιστεί και να είμαστε ταυτόχρονα ικανοί να το υλοποιήσουμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Στη συνέχεια θα λάβει τον λόγο ο κύριος Μαρινέσκου. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συγητές συναδέλφους για τη συνεργασία και για την σκληρή δουλειά που κάναμε μαζί. Ευχαριστώ και τον κύριο Σασόλη για τις δύο εκθέσεις, γιατί τώρα είναι συμπληρωματικές και είχαμε μια αγαστή συνεργασία. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να αναφερθώ στην Κομισιόν και να πω ότι με την διαγραφή της υποχρεωτικής, του υποχρεωτού διαχωρισμού των υπηρεσιών δεν έχει μειωθεί ο αντίκτυπος αυτής της έκθεσης. Δεν μπορούσαμε να στηρίξουμε αυτή την πρόταση διότι από τεχνική άποψης ήταν πάρα πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί. Επίσης, άποψή μας είναι ότι η μείωση του κόστους δεν γίνεται μέσω αυτού του διαχωρισμού, αλλά με άμεσες διαδρομές, αεροδιαδρόμους και μια αρχιτεκτονική του χώρου που θα μειώσει τον χρόνο πτήσης. Όπως είδατε, ε, στους προλαλήσαντες αυτή η κατάσταση αντανακλάται. Υπάρχει μια επιφύλαξη ανάμεσα στα κράτη-μέλη, ένας φόβος για τους, τις θέσεις απασχόλησης και για την, ε, την διοίκηση γενικά, την ανεξαρτησία των εθνικών αρχών. Αυτή η ανεξαρτησία είναι ένα συν για την ασφάλεια της αεροπορίας και για όλη την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων σε αυτό τον τομέα. Εμείς στη Ρουμανία λέμε από αυτό που φοβάσαι δεν γλιτώνεις. Είμαι βέβαιος ότι στο τέλος ο ενίος ευρωπαϊκός ουρανός θα μείνει εκεί που είναι η θέση του προς όφελος όλων των εμπλεκομένων φορέων αυτού του κλάδου και προς όφελος κυρίως των επιβατών που είναι, είναι οι δικαιούχοι και οι χρήστες αυτής της υπηρεσία. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Τώρα στη συνέχεια θα λάβει τον λόγο ο κύριος Σασόλη, παρακαλώ. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος γιατί μακρηγόρησα στην πρώτη μου παρέμβαση. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τον κύριο Μαρινέσκου και να σας πω ότι μιλάμε για επιτήρηση, για πάυση των συνθήκων κατακαιρματισμού και ότι θα πρέπει τελικά να έχουμε αυτή τη στιγμή έναν ευρωπαϊκό οργανισμό ενέργεια κυκλοφορία που θα βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ασφάλεια. Ο κύριο Φεραίρα, πώ μα λέει ότι θα διηγηθούμε σε χαμηλότερο επίπεδο ασφάλεια. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Σα καλώ όλου σα να διαβάσετε τα δύο αυτά κείμενα, τι δύο εκθέσει, προκειμένου πραγματικά να συνειδητοποιήσετε ποιε είναι οι δυνατότητε που έχουμε και αν πραγματικά όντω μιλάμε για διδικοποίηση. Εμεί σε κανένα σημείο δεν μιλάμε για διδικοποίηση. Κυρία Επίτροπε, όσον αφορά τι ε, κατεξοδότηση πράξη, ξέρετε ότι υπάρχει σαφή τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υπερβαίνει ουσιαστικά τι ε, επιμέρους επιτροπές. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να μπορεί να ελέγχει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αύριο θα ψηφίσουμε τι δύο αυτέ εκθέσει από κοινού θα έχουμε στο μέλλον πάρα πολλή δουλειά να επιτελέσουμε στο μέλλον, τουλάχιστον για να πείσουμε το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Σασόλη. Ολοκληρώσαμε τώρα με αυτή τη συζήτηση το θέμα και θα ψηφίσουμε αύριο στις 12 το μεσημέρι. Και έτσι περνάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι η έκθεση του κ. Μάγερ για τα οργανωμένα ταξίδια και ταξιδιωτικά πακέτα και εξατομικευμένα θέματα ταξιδιωτικών διακανονισμών. Ο κύριος Μάγερ, τέσσερα λεπτά πρώτος παρακαλώ.